Kolleginnen und darf Sie zur Fortsetzung unserer Tagesordnung. Κυρίες και κύριοι, ε, συνεχίζουμε λοιπόν τις ε, εργασίες μας και πρέπει να σας πω χαίρομαι πολύ που έχουμε κοντά μας την Αντιπρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα τη εκπρόσωπο. Και χαίρομαι επίσης που θα ακολουθήσει η συζήτηση. Νομίζω ότι τις ερωτήσεις μας θα πρέπει ε, κάπως ε, να τις ε, εστιάσουμε στο τι ακριβώς συνέβη εχθές στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων Ουκρανία, Συρία και να μην ρωτήσουμε τα πάντα επί του επιστητού. Και Ίσως θα μπορούσα και εγώ να πω κάτι από το τελευταίο μου ταξίδι. Καλύτερα όμως να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, σε αυτά που είναι επίκαιρα. Ε, η Ντόρις ήθελε να είναι παρούσα στη συζήτηση για τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Θα ήθελα λοιπόν, συνάδελφοι, να, είσαστε, να επιδείξετε λιγάκι συνέπεια, έτσι ώστε να έχουμε και μια συνεπή συζήτηση, συνεκτική περισσότερο. Κάθι, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά ξανάρχομαι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θεωρώ θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να σα δώσω μια επισκόπηση των θεμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων χτε που αντιμετώπισε πολλά σημαντικά θέματα. Βέβαια θα με ενδιαφέρει να ξέρω ποια είναι τα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν εσάς ιδιαίτερα και να εξασφαλίσω ότι θα έχετε τι κατάλληλε απαντήσεις. Ας ξεκινήσω όμω με τη Βοσνία Ζεγοβίνη όπω είπε και ο πρόεδρο σα. Έτυξε αυτό το θέμα στην εισαγωγή μου προς το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Αυτό το οποίο μας εντυπωσίασε όλους είναι ότι αυτές οι βίες διαδηλώσεις προέρχονται από τη ματέωση κυρίως που νιώθει ο πληθυσμό λόγω της οικονομικής κατάστασης στη Βοσνία Ρεσεγοβίνη. Όσοι παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση ξέρουν ότι η ανεργία έχει φτάσει στο 45% περίπου. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των νέων ανέργων και ενώ δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη βία σε οποιοδήποτε πλαίσιο, σε οποιασδήποτε περιπτώσει, είναι φανερό ότι χρειάζεται πραγματική ηγετική ικανότητα από τους ηγέτες της Βοσνίας Ζεγοβίνη. όλοι αυτοί που έχουν δει την κατάσταση όχι μονάχα στο Σαράγεβο αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, χρειάζεται να υπάρξουν ηγέτες οι οποίοι θα προχωρήσουν τη χώρα. Μα δείτε τι γίνεται σε αυτή την περιοχή, θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος που γίνεται γενικά στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά την απάντηση, την ανταπόκριση στις ανάγκες πολιτικές και οικονομικές ανάγκες του λαού, αλλά φαίνεται ότι δεν προχωρά η Βοσνία Ζεγοβίνη. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από ό,τι οφόρο τιμής στο συνάδελφο μου, στον Στέφεν Χιούλε, ο οποίος έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Και συνεχίζονται οι προσπάθειες ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ υπηρεσιών της Κομισιόν, μαζί με τους εταίρους μας από την άλλη οχθή του Ατλαντικού για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια πραγματική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωση εκεί. Παίζουμε ένα ηγετικό ρόλο σε επίπεδο περιφερειακό, αλλά πρέπει να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. <clears throat> Αναφερθήκαμε και στην πρόσφατη διάσκεψη κορφής με τη Ρωσία και έκανα μια σύντομη επισκόπηση. Δεν ήταν business as usual. Είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον πρόεδρο Πούτιν, κύριο για τη γειτονιά μας. Αντιμετωπιστήκαν οι διαφορές με ένα ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο σε τριμερείς συναντήσεις μεταξύ των τριών πρόεδρων που κάθισαν μαζί και συζήτησαν ανοιχτά όλα αυτά τα θέματα και στη συνέχεια σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δώσαμε ένα σαφές μήνυμα σε σχέση με τις ανησυχίες μας ο Ρώσος Πρόεδρος και η δική του πλευρά ανέφεραν τις δικές τους ανησυχίες και όλο αυτό οδήγησε σε διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η επίπτωση ορισμένων από τις συμφωνίες μας, ιδίως η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Ρωσίας με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, πώς αυτά επηρεάζουν και ευνοούν την οικονομία της Ρωσίας και πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση η οποία έχει δημιουργηθεί. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε λοιπόν να ανοίξουμε το δρόμο για νέες συμφωνίε στο μέλλον. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι καλή η διμερή μα σχέση με τη Ρωσία, αλλά πρέπει να είναι μια σχέση που να βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό για την κατεύθυνση που ακολουθεί κάθε πλευρά και για την καλύτερη κατανόηση από τη ρωσική πλευρά του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τρόπου με τον οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε τη σχέση μας με κυρίαρχα κράτη στην περιοχή αυτή. Για το κύριο μέρος τώρα του Συμβουλίου Υπουργών είχαμε μια μακρά συζήτηση για την ανατολική εταιρική σχέση, μια, ένα απολογισμό τι έγινε στη συνάντηση του Βίλνιους, τι έγινε στην Ουκρανία. Κύριε Πρόεδρε και εγώ ήμουνα στην Ουκρανία όπως και εσείς. Ο Επίτροπος Φιούλε και άλλοι θα μεταβούν στην Ουκρανία. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να πούμε για την Ουκρανία. Και στο πλαίσιο <clears throat> της προσπάθεια μας μετά τη διάσκεψη του Βίλνιους μας ενδιαφέρει να υποστηρίξουμε τη Μολδαβία και τη Γεωργία με φιλοδοξία να υπογράψουμε συμφωνίες με αυτές τις χώρες πριν από το τέλος της θητείας της τρέχουσας Κομισιόν. Έχουμε αντλήσει ορισμένα διδάγματα από τη διάσκεψη του Βίλνιους, τη σημασία να κατήσουμε πολιτική παρουσία στο πιο ψηλό επίπεδο, όπως προχωρούμε προς την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ρήγα. Θέλουμε να υπάρξει η ετοιμότητα των Υπουργών για να κάνουν επισκέψεις υψηλού επίπεδου και προσωπικά και ομαδικά υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές δεν έχουν ακολουθήσει πάντα οι Υπουργοί αυτή την οδό αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να διευρύνουμε και την συμμετοχή μας και την επαφή μας με διάφορες ομάδες της κοινωνίας και για να διαλύσουμε τις παρεξηγήσεις σε σχέση με τη μορφή αυτής της συμφωνίας, αυτό είναι πολύ σημαντικό στη Μολδαβία. Αυτό σημαίνει όμως και οι κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και προσβλέπω προς την υποστήριξή σας αυτού του έργου σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Έχετε καταφέρει να πλησιάσει όχι μονάχα τα κοινοβούλια, αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Επίση, πρέπει να υπάρξει επαφή και μεταξύ επιχειρηματιών και τοπικών αρχών, ώστε να γίνει κατανοητό από τι χώρε αυτέ το τι δυναμικό μπορεί να απελευθερωθεί από αυτέ τι συμφωνίε και πώ μπορούν να βοηθηθούν οι επιχειρήσει του και η κοινωνία του ω σύνολο. Τα μηνύματα αυτά λοιπόν θα πρέπει να διαδοθούν και από τις αντιπροσωπείες μας με μια δημόσια διπλωματία για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και να εξασφαλίσουμε ότι ο διάλογος με τη Ρωσία θα γίνει πιο εντατικός. Αναφερθήκαμε στην επίσκεψη που έκανα στην Ουκρανία δύο φορές τις τελευταίες δέκα μέρες. Έχω πάει εκεί. Πραγματικά είναι ανησυχητικά τα πράγματα, τα είπα σε όλες τις συνεντεύξεις τύπου. Εγώ εντυπωσιάστηκα για την αλλαγή που έχει γίνει από τον Νοέμβριο στην πρώτη μου ε, επίσκεψη και την πρόσφατη επίσκεψή μου. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ένταση, πολύ μεγαλύτερη αστυνομική παρουσία Τώρα έχουν κάπως καλμάρει τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι όλοι έχετε παρακολουθήσει τι έχει γίνει, πόσα θύματα υπήρξαν από αυτή τη βία και έχετε ακούσει ιστορίες και αφηγήσει από πολλούς που ήταν παρόντες εκεί. Είναι πολύ σαφές επίσης, άμα δείτε, τη βία που ασκείται στην Ουκρανία, ότι <clears throat> δεν υπάρχει τίποτα προς την κατεύθυνση μιας ανεξάρτητης έρευνας που στον 20ο αιώνα θα θέλαμε να γίνεται σε μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αδικοπραγούντες θα έλθουν ενώπιον της δικαιοσύνης και κάτι το οποίο είναι σαφές είναι ότι είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να δώσει αυτό το μήνυμα ότι θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε εμπειρογνωμοσύνη, διαμεσολάβηση, υποστήριξη κάθε είδους σε όλα τα επίπεδα με οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, με τους εμπειρογνώμονές μας. Μπορούμε να βρούμε σε κάθε επίπεδο τα απαραίτητα άτομα. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να βγει αυτή η διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχουμε κάνει σαφώς αυτή την προσφορά προς την Ουκρανία. Επίσης, και ξέρω ότι και εσείς κύριε Πρόεδρε ενεπλάκητε ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη συζητήση για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και της ανάγκης να μην γυρίσουμε όχι μόνο στο Σύνταγμα του 2004, αλλά σε ένα Σύνταγμα του 2004 συν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα στοιχεία από αυτό το Σύνταγμα, αλλά να αφαιρέσουμε αυτά τα οποία ε, να αφαιρέσουμε αυτά που δίνουν υπερβολικές εξουσίες στους ε, ανακριτές δικαστές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να δράσουμε και σε άμεσο επίπεδο, βραχυπρόθεσμο, για να αντιμετωπίσουμε τις ε, αναταραχές και τις ανησυχίες που έχει ο πληθυσμός που διαδηλώνει στο ΜΕΙΔΑΝ, αλλά και τις πιο μακροχρόνιες πτυχές, ώστε στο τέλος το Σύνταγμα της Ουκρανίας να είναι πιο επαναξισορροπημένο και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισορροπία των εξουσιών. Είναι μια διαδικασία που την έχουμε υποστηρίξει. Βλέπουμε την νομοθεσία περί αμνηστίας. Υπήρχαν τέσσερις επιλογές. Αυτή που διάλεξε το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ήταν αυτή που διάλεξε. Και υπάρχουν τώρα και κάποιες καταληκτικές προθεσμίες και φυσικά μας ενδιαφέρουν οι καθαρές και αμερόληπτες εκλογές στο τέλος της διαδικασίας, ώστε όλοι να μπορέσουν να κάνουν τη φωνή τους ακουστή σε αυτές τις εκλογές. Είχα επίσης επαφές, όπως ξέρετε, και σε σχέση με τα οικονομικά θέματα. Όταν πήγα τον Νοέμβριο, μίλησα για 3,5 ώρες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να δείξω όλες τις πτυχές των οικονομικών προβλημάτων της χώρας, βράχη πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και σε όλες τις συζητήσεις που είχα με τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και τις επιχειρηματικές δομές της χώρας. Τόνισα ότι υπάρχει από τη δική μας πλευρά η θέληση να υποστηρίξουμε τις προκλήσεις που έχει ενώπιον της η Ουκρανία. Αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς μεταρρυθμίσεις. Μόνο αν θέλουν να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να προχωρήσει η χώρα τους. Πρόκειται για μια αναδιοργάνωση της βιομηχανίας για να γίνει πιο ανταγωνιστική να αντιμετωπιστούν τα βραχυχρόνια, τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα με το έλλειμμα του προπολογισμού κτλ. Και την Πέμπτη θα πάω στη Ουάσιγκτον να συναντήσω την Κριστή Λαγκάρτ. Και ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι η Ουκρανία. Αλλά και η Μολδαβία και η Γεωργία είναι πάρα πολύ σημαντικέ Έχουμε πολλές ε, ανάγκες να προωθήσουμε όλα αυτά τα θέματα προς την υπογραφή συμφωνιών και επίσης την υποστήριξή μας εάν υποστούν πιέσεις για, την, ε, για να εμποδιστεί η συμφωνία της συμφωνίας DCFTA. Και έχω τονίσει σε όλους αυτούς τι σημαίνει αυτό για τους λαούς τους, για τις κυβερνήσεις τους, ποιες ευκαιρίες ανοίγονται ενώπιόν τους. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες προς τις χώρες αυτές σε τακτική βάση. Οι Υπουργοί ήθελαν επίσης να συζητήσουν και διάφορα σημεία ε, τα οποία αφορούν την νότια γειτονία. Στα πλαίσια των ε, περιφερειακών προκλήσεων δεν θα εκπλαγείτε βεβαίως ε, εάν σας πω ότι η σκέψη τους αναφέρθηκε στο Ιράκ, ε, στην ε, κατάσταση η οποία πλέον μας απασχολεί ιδιαιτέρως. Πρέπει να πω ότι ήταν ιδιαίτερη και η χαρά των εκπροσώπων της χώρας αυτής στις διεθνείς διαδικασίες. Μας απασχολεί όμως πάρα πολύ, μας απασχολούν τα όσα συμβαίνουν στο Ιράκ επίσης ο Λαχτάρ Μπραχήμι όσον αφορά τη Συρία συνεχίζει ε, την ε, εργασία του, συζητήσεις ε, με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης αλλά και του καθεστώτος. Θα θυμάστε ότι ήμουν και στη Γενέβη 1 και στη Γενέβη 2. Είναι σαφές ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση από πλευρά της διεθνούς κοινότητας, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα αλλά είναι εξίσου σαφές ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχει έλλειψη ε, κατανόησης ε, σχετικά με το τι πρέπει να γίνει εφ' εξής. Ε, συζητούμε με τον Λακτάρ Μπραχίμη ε, γιατί η εργασία την οποία έχει αναλάβει είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, η θέση των Συρίων γυναικών επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρή. Οποιουδήποτε δόγματος, οποιασδήποτε ομολογίας θα πρέπει, θέλουν και αυτές να συζητήσουν έτσι ώστε να προωθηθεί η ειρήνη. Κρίμα, και ντροπή γιατί ήταν πάρα πολύ λίγες οι γυναίκες στη επί στην αίθουσα των ε, συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων. Ε, Υπήρχαν ορισμένες γυναίκες, αλλά πάρα πολύ λίγες στις αντιπροσωπείες και από τις δύο πλευρές. Ε, βεβαίως, ε, οι ε, γυναίκες με τις οποίες ήρθα σε επαφή πραγματικά έχουν διάθεση να δουλέψουν, θέλουν να παίξουν μεγαλύτερο, σπουδαιότερο ρόλο στο μέλλον. Επίσης, συζητούμε με τα κράτη-μέλη υπό το ε, Λουξεμβούργο για τα σχετικά με το Συμβούλιο Ασφαλείας όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια η οποία θα χρειαστεί κάποια στιγμή παρακολουθούμε τις δυσκολίες οι οποίες ε, ε, ε, υπάρχουν στη Νέα Υόρκη σχετικά με ένα ενδεχόμενο ψήφισμα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να προωθηθεί η βοήθεια επιτόπου στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι παγωμένα κονδύλια θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή του χημικού ε, και το Λίβανο μας απασχολεί. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε μια πραγματική αποτελεσματική κυβέρνηση. Ε, έχουμε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό επανειλημμένα. Τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες ε, ημέρες ε, ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και εν ώψη και των εκλογών. Αλλά βεβαίως 25% και πάνω του πληθυσμού αποτελείται από πρόσφυγες, πράγμα που κάνει τον πληθυσμό αυτό εξαιρετικά ευάλωτο. Είναι πάρα πολύ ε, τρωτή η κατάσταση και βεβαίως ε, τα διακυβεύματα και οι προσκλήσεις πάρα πολύ μεγάλα τρίτη επέτειος, τρίτο γενέθλιο της ε, από την ε, από την εξέγερση στην Αίγυπτο. Πολλά έχουν γίνει, πολλοί σε κόσμος έχει βρεθεί στις φυλακές ενώ δεν θα έπρεπε. Μας απασχολεί αυτό, αλλά μας απασχολεί εξίσου και η ολοένα αυξανόμενη βία ε, και οι αυξανόμενες τρομοκρατικές ε, ενέργειες. Γνωρίζουμε ότι και στην Αίγυπτο και στις γειτονικές ε, περιοχές υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ θα ήθελα δεν να σημειώσω την εξαίρετη εργασία του Σταύρου Λαμπρινίδη όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και οπωσδήποτε πρέπει να συζητήσουμε και την κατάσταση και στην Τινησία αλλά και στη Λιβύη. Στη Λιβύη μας απασχολεί πάρα πολύ όλο αυτό το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί ε, και το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ, ε, κενό εξουσίας στην ε, ε, γειτονική κατάσταση, στις γειτονικές περιοχές επίσης ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στην Ιεμένη. Ξέρουμε ότι υπάρχει δυνατότητα διαλόγου, δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, ιδιαίτερα ευαίσθητες χώρες να προχωρήσουν παρόλα αυτά μπροστά. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να βελτιωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις. Να σας πω και δύο λόγια κύριε Πρόεδρε όσον αφορά την ε, Κεντρική Αφρική. Ε, έχουμε ε, συναντηθεί με τον στρατηγό Φιλίπ Ποντιέ, ο οποίος είναι γενικός υπεύθυνος των επιχειρήσεων εκεί και ξέρουμε ότι, την, ότι η κατάσταση μπορεί να προχωρήσει. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Βαρόνι Άστον. Ξέρετε, τώρα έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί 25 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Και κανονικά, ε, ακόμα και αν ε, έφευγε τώρα η κυρία Άστον, μόνο για τις ερωτήσεις θα εξαντλείται ο χρόνος και δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε τις απαντήσεις. Άρα ερωτώ οι συντονιστές να πάρουν δύο λεπτά και οι υπόλοιποι να είναι πολύ πιο σύντομοι. Αν συμφωνείτε να δούμε τι θα κάνουμε, μέχρι πού θα προχωρήσουμε. Θα προσπαθήσω να μοιράσω το χρόνο στις ε, πολιτικές ομάδες, αλλά ξέρετε δεν έχει νόημα να γίνονται ερωτήσει και μετά να μην υπάρχει χρόνος για τις ε, απαντήσεις και ούτε είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνονται οι ίδιες και οι ίδιες ε, ερωτήσεις. Αν το κάνουμε αυτό θα κερδίσουμε χρόνο. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος ερωτήσεων, ο κύριος Σαλαφράνκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήλθατε κυρία Αστόν. μα λείπατε που δεν σα είχαμε δει τόσο καιρό. Τρία θέματα. Πρώτα η Ουκρανία. Παρά τι επικρίσει που ακούσαμε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή μα, νομίζω ότι η δική σα παρουσία αυτή του κυρίου Φίλε και των μελών του Κοινοβουλίου δίνει πρόσθετε εγγύησεις για την ασφάλεια των αντιφρονούντων, τη αντιπολίτευση και των διαδηλωτών. Νομίζω ότι μετά από την κατάργηση των περιοριστικών της ελευθερίας νόμων, και της έγκρισης του νόμου περί αμνηστίας, υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης που επιτρέπει να υπάρξει ένας ορικός χάρτης για, και για μια νέα κυβέρνηση και για μια συνταγματική μεταρρύθμιση και επίσης για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια διαδικασία για πρόορες βουλευτικές ή προεδρικές εκλογές που θα δώσουν μια ειρηνική διέξοδο στην, ε, στις διεκδίκησεις του λαού. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω για την Ουκρανία είναι αν θεωρείτε το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περάσει από τη διευκόλυνση στην διαμεσολάβηση για να μπορέσει και να υπάρξει κάποιος φορέας που θα ελέγξει ότι τηρούνται τα υπεσχημένα. Αναφερθήκατε και στη συνάντησή σας με την κυρία Λαγκάρτ στο Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω αν ε, η κυρία Λάγκαρτ θα πει και καμιά κουβέντα στην κυρία Νιούλαντ μετά από την πρόσφατη στιχομηθεία που ξέφυγε από τα χείλη της κυρίας Νιούλαντ. Επίσης, σε σχέση με την Ελβετία. Τι γίνεται μετά το δημοψήφισμα. Αυτό είναι μια απόφαση που μπορεί να αφορά ένα εκατομμύριο πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτεστε να αναστείλετε τις συμφωνίες οι οποίες ισχύουν αυτή τη στιγμή ή ένα πάγωμα των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση των θεσμικών σχέσεων. Τελευταίο ερώτημα, η Κούβα. Θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι η συμφωνία που έχετε πετύχει στο Συμβούλιο είναι μια συμφωνία τρίτης γενιάς που βασίζεται και στη δημοκρατική ρήτρα και στην κοινή θέση του Συμβουλίου που εξακολουθεί να ισχύει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε κυρία Αστόν. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ε, για το ρόλο των γυναικών και ελπίζω στην ε, Γενέβη 3 να υπάρχουν γυναίκες στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Στην Ουκρανία όταν την επισκεφτήκαμε πραγματικά εντυπωσιάστηκα εκεί από ε, τον ενθουσιασμό, τη μαχητικότητα των γυναικών στην πλατεία Μαϊντάν και κυρίως από το ότι οι γυναίκες απευθύνονται σε εμά και μας καλούσαν να χρησιμοποιήσουμε την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όχι μόνο γιατί αυτό θα πειράσει τους ίδιους, αλλά στη τελική ανάλυση κάτι τέτοιο δεν είναι και προς δικό μας όφελος ε, γιατί επ' αυτού έχουμε δει να υπάρχουν αντιφατικές τοποθετήσεις κατόπιν για την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία από το Δεκέμβριο του 2012 ε, υπάρχουν εκτοξεύτηκαν απειλές που τελικά υλοποιήθηκαν για το γενοκτονία και από το Μάρτιο του 2013 ε, πολλοί ζητούν ζητάνε ή λένε ότι επιτόπου αυτό το λένε οι ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις ότι θα υπάρξει στρατός επιτόπου. Ε, αυτό πότε όμως θα υπάρξει ε, μετά τη γενοκτονία. Και κατόπιν η Λιβύη, τελευταίο ερώτημα. Βλέπω να υπάρχει μόνο μία πολύ μικρή γραμμή στις δηλώσεις σας ότι αυτό συζητήθηκε. Ε, είπατε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν οι κυρώσεις. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα κράτη-μέλη και να τα ε, καλέσετε για τις ευθύνες τους, για το τι διαδραματίζεται στη Λιβύη, γιατί φέρουν ευθύνη, διότι δεν προχωρούν ε, στο συντονισμό, αρνούνται το συντονισμό υπό την καθοδήγησή σας. Σας ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρο. Βαρόνι σας καλωσορίζουμε και σας ε, ευχαριστούμε πολύ για την περιεκτική ενημέρωσή σας σχετικά με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα χθες. Διάβασα τα συμπεράσματα και εντυπωσιάζομαι από το ότι στο κείμενο δεν λέγονται πολλά για τη Συρία και δεν μπορώ να φανταστώ ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Το γεγονός λοιπόν ότι στο κείμενο περιλαμβάνονται τόσο λίγα λόγια, αυτό για μένα σημαίνει ότι όλα είναι ρευστά και ότι είναι πολύ δύσκολο να διατυπωθεί μια θέση. Θα ήθελα να ε, μου πείτε αν έχω δίκιο. Δεύτερον, όσον αφορά τη Ρωσία, διάβασα σε ένα άρθρο στο γαλλικό περιοδικό Express την προηγούμενη εβδομάδα ότι από ό,τι φαίνεται ο κύριος Σούβανοφ ε, σας είπε ότι η Ρωσία προτίθεται να ε, συστήσει και αυτή στη δική της γεωγραφική πλευρά ένα είδος ένωσης. Ισχύει αυτό, μπορείτε να μας ενημερώσετε παρακαλώ επ' αυτού. Και τέλος και εγώ θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον όσον αφορά στην Ουκρανία, γιατί από τη μια μας λέτε ότι θα μιλήσετε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να δείτε τι είδου πακέτο μπορεί να χορηγηθεί στη χώρα αυτή, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ε, κατά πόσον υπάρχει και το ενδεχόμενο των κυρώσεων. Κυρώσεις στην περίπτωση κατά την οποία επιδεινωθεί η κατάσταση. Και τέλος και κάτι άλλο. Μπορείτε να μας πείτε την ε, σχετικά τη δική σας θέση για αυτή την ατυχέστατη έκφραση που εξεστόμησε η κυρία Γιούλαν τη ε, Αμερικανίδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε κρίσιμη χρονική στιγμή και για τις σχέσεις μας ε, με τη Ρωσία και με τις ε, χώρες της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, πιο συγκεκριμένα σχετικά με τη διαμεσολάβηση Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι σε θέση να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή σε αυτή τη διένεξη και αυτό το ρόλο της τον αναγνωρίζουν και οι δύο πλευρές. Και κάτι άλλο σχετικά με τα συμπεράσματα εχθές του Συμβουλίου για την Ουκρανία. Στο τέλος των συμπερασμάτων αναφέρεται ότι η Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία, δεν θυμάμαι ακριβώ τη διατύπωση, αλλά κάπως ε, από ό,τι κατάλαβα είναι ότι δεν τελειώνει εκεί η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, Ουκρανία. Και θέλω να μου πείτε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς το ερμηνεύουν οι ίδιοι Ουκρανοί και επ' αυτής της ε, διατύπωσης υπήρξε συνένεση και κάτι σχετικά με την Βοσνία. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε έτσι ώστε να παρεμποδίσει τα πολιτικά κόμματα να δώσουν μια αδιαμφισβήτητη εθνοτική χρειά στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα αυτή. Συγγνώμη τον κύριο Δόκτωρα Κέρκο, ο οποίο έπρεπε να γυρίσει στο Λονδίνο. Θέλω να θίξω ένα θέμα που δεν έχει αναφερθεί. Παλαιστίνη και Ισραήλ, ιδίω σε αυτή τη στιγμή υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στο Ισραήλ γιατί φαίνεται να υπάρχει μια ε, νοοτροπία οχύρωσης από την πλευρά του Ισραήλ, γιατί βλέπουν ότι δεν γίνεται καμία πρόοδο σε σχέση με τα θέματα της Παλαιστίνης. Μπορείτε να μας πείτε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, αν βλέπετε να υπάρχει κάποια πρόοδο μετά την παρέμβαση του κυρίου Κέρι. Δεν θα ήθελα να πω ότι είναι αντισημητικό αυτό, αλλά κάπως τους έχει πατήσει στον κάλο και αυτό φαίνεται να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Έχετε την ε, κάποια άποψη αν τελικά οι θρησκευτικέ ε, τα θρησκευτικά κόμματα είναι αυτά τα οποία κινούν τα νήματα ή αν δεν έχουν καμία δυνατότητα να προχωρήσουν τα πράγματα. Και ε, ε έχω ανησυχίες για τις ε, την περίπτωση των Βεντουίνων και του οικισμού στην περιοχή ε1 που είναι τεράστιες και προκαταλαμβάνουν ενδεχομένω και τις λύσεις. Και νομίζω ότι δεν πρόκειται να ξαναβρεθούμε ίσως εύκολα όπως είμαστε τώρα σε αυτή την Επιτροπή. Είχαμε τις πολιτικές μας διαφορές, αλλά θέλω να σας συγχαρώ για το ότι παίξατε πολύ καλά με ένα δύσκολο χέρι χαρτιών και καταφέρατε να πετύχετε πολλά πράγματα παρά τις δυσχέρειες που είχατε και έχετε απόλυτα την ε, σωστή μου αξιολόγηση τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Άστον για την έκθεσή της. Θα ήθελα να σταθώ μόνο σε δύο σημεία της ε, εκτενούς παρέμβασής σας για την Ουκρανία. Η πολιτική μου ομάδα κρατάει μια σαφή θέση. Μόνο ο λαός της Ουκρανίας θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του, χωρίς κυδαιμονίας, χωρίς παρεμβάσεις από κανένα. Ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε. Δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> θέλει να παίξει το ρόλο του, κυδαιμόνα του κυδεμόνα και εμπλέκεται σε μια υπόθεση που δεν, της, ε, που δεν είναι δική της υπόθεση. Ούτε και η Ρωσική Ομοσπονδία φυσικά πρέπει να παρέμβει, ανεξάρτητα από τις γεωστατηγικές επιδιώξεις. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία πίεση, καμία κυδαιμονία. Είδαμε τη βία που ασκήθηκε στους δρόμους. Μα και σε πολλά κράτη-μέλη υπήρξε βία. Στη χώρα μου, στην Ισπανία, υπήρξαν αυτοί οι διαδηλωτέ που βρέθηκαν γύρω από, το, τα κόρτες και αντιμετώπισαν τα ΜΑΤ. Και βγήκε ένας νόμος για να περικόψει το δικαίωμα του διαδηλώνει. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα εναντίον των ε, διαδηλωτών στην πλατεία Ποσειδόνος στη Μαδρίτη. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μοναδικό γεγονός. Επομένως και αυτά που γίνονται στην Ουκρανία δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εμείς δεν συμφωνούμε για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε εμείς κάποιοι οι οποίοι μπορούμε να δώσουμε μαθήματα σε κάποιους άλλους και να τους κυδεμονεύσουμε. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο ρόλο. Και δεν πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρήσουν ότι πρέπει να δώσουν μαθήματα στην Ουκρανία. όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, να μπούμε όπου, εκεί που υπάρχουν διαδηλώσει, τότε πηγαίνετε από την Αθήνα, πηγαίνετε από την Πορτογαλία, πηγαίνετε από τη Μαδρίτη, όπου υπάρχουν διαδηλώσει, κάντε κάτι. Μα τι πρέπει να κάνει κανεί, πρέπει να χρησιμοποιήσει την νομοθεσία, πρέπει να ζητήσει από το κάθε κράτο να λύσει τα εσωτερικά του προβλήματα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω δύο λόγια ε, από την σκοπιά της Επιτροπής, Υποεπιτροπής Άμυνας ε, για την ε, Κεντρική Αφρική και εγώ ε, έχω τον ίδιο προβληματισμό με την συνάλφα Άννα Γκόμες. Ε, μιλάμε πολύ καιρό ε, για αυτήν την αποστολή. Ποιες είναι οι δυνατότητες, τα ενδεχόμενα να υπάρξει αποστολή δυνάμεων σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνα της Γαλλίας μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Έχει αναφερθεί στις 21 Φεβρουαρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει πού βρισκόμαστε σε σχέση με τους 500 υπεσχημένους ε, στρατιώτες. Επίσης, ε, Λιβύη, όπως είπε και η Άννα, εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε μία ε, αποστολή ε, e SDC για την, στην χώρα αυτή. Μαθαίνουμε πάντως ότι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, τουλάχιστον αυτό διαρρέει στον τύπο, κάνουν κάποιες μεμονωμένες, μονομερείς προσπάθειες ε, να βοηθήσουν στην ανασύσταση ε, στρατιωτικών σχηματισμών στην Λιβύη. Δεν έχουμε όμως θεσμική ε, δυνατότητα ή νομιμοποίηση ή εντολή έτσι ώστε να κάνουμε από κοινού τέτοιες προσπάθειες. Η κάθε χώρα είναι μόνη της. Για τη Λιβύη όμως δεν κάνουμε τίποτα. Και τέλος για την Βοσνία υπενθυμίσατε και εδώ ότι έχουμε σημαντικό σημαντικό, ε, ε, ένα σημαντικό πολιτικό οπλοστάσιο στην χώρα αυτή, αλλά έχουμε όμως και στρατιωτικό. Ε, αλλά πρέπει να πω ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή στην Βοσνία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της αποστολής που τίποτα δεν μπορεί να κάνει απέναντι στους οικονομικούς και κοινωνικούς κλειδονισμούς στους οποίους αντιμετωπίζει η χώρα αυτή. Σας ε, ευχαριστώ πολύ ε, για τις ερωτήσεις. Κύριε Σαλαφράγκα, και εσείς μου λείψατε. Ε, ξέρετε, όμως ήμουν πολύ απασχολημένη την τελευταία, τον τελευταίο καιρό. Σχετικά με την Ουκρανία, μία από τις ερωτήσεις σας και τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει ως προς την διαμεσολάβηση ή διευκόλυνση των ε, σχέσεων. Αυτό που είπαμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, στον πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στην κοινωνία των πολιτών είναι ότι εμείς ε, δεν θα παρέμβουμε, αλλά με μεγάλη μας χαρά να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε με όποιον τρόπο κριθεί κατάλληλος. Και όσον αφορά ε, το τι μπορούμε να κάνουμε εξαρτάται από το που θα μας ζητήσουν να βοηθήσουμε. Από εκεί θα εξαρτηθεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πει κανείς ότι εντάξει ε, θα ε, διαμεσολαβήσουμε. Αλλά από ό,τι ξέρετε και από ό,τι γνωρίζω και εγώ από την εμπειρία μου, η διαμεσολάβηση μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και ε, είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρει κανείς ότι θα κάνει αυτό το οποίο είναι χρήσιμο. Και αυτό όμως πρέπει οι ίδιοι να το συμφωνήσουν έτσι ώστε να μην παρέμβουμε αδικαιολόγητα. Όμως είναι αλήθεια ότι μας έχει γίνει πρόταση σχετικά με την κύρια Γιούλαντ. Να σας πω κάτι, ήταν μια ιδιωτική συζήτηση. Κάποιος το έβαλε στο YouTube ε, και εντάξει δεν θέλω να πω τίποτα άλλο από αυτού. Εντάξει, ο καθένας ε, λέει ό,τι θέλει αν θέλετε στις ιδιωτικέ της κατηδίαν συζητήσεις. Δικαίωμά του είναι. Τώρα για την Ελβετία. Έχουν περάσει, ή μάλλον θα περάσουν τρία χρόνια για να αποφασίσει η κυβέρνηση το τι θα κάνει και από ό,τι κατάλαβα ε, θα καταθέσουν μια πράσινη βίβλο σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του δημοψηφίσματος. Και τώρα ε, η Επιτροπή και εμείς ε, εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τη συνθήκη της Λισαβόνας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον και για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η απόφαση αυτή για πάρα πολλές ε, συμφωνίες που έχουμε συνάψει με την Ελβετία. Όπως ξέρετε πολύ καλά, οι σημαντικοί παίκτες και τα μεγάλα κόμματα δεν ήταν εκείνοι που ζήτησαν το δημοψήφισμα, γι' αυτό πρέπει να δούνε τι θα κάνουν. Πάντως η ελευθερία κινήσεων είναι πυλώνας των, των σχέσεών μας, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστική σημασία σχετικά με τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Και ελπίζω να ε, ξεβρεθεί μια ικανοποιητική λύση που ε, να είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Σχετικά, Ούβα, σωστά είπατε, αυτά τα οποία γίνονται είναι σωστά, ο τύπος είναι θετικός, αρκετά θετικός στην Κούβα και νομίζω ότι τελικά παραμένουν και εμείς παραμένουμε πιστοί στις υποχρώσεις μας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω όμως ότι η λύση είναι καλή, είναι εξάλλου μια ομόφωνη απόφαση, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Κυρία Γκόμες, ε, συμφωνώ όπω πολύ καλά γνωρίζετε με τη θέση σας ε, σχετικά με τις γυναίκες. Είχαμε πάρα πολλέ συζητήσει ε, και με και χωρίς την Ουκρανία για το τι πρέπει να γίνει για να ασκηθεί πίεση αλλά και για να προσφέρουμε υποστήριξη αυτή η δυτή προσέγγιση που έχουμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις με τα κρατη με, τους, τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά τις δυνατότητες, ε, τις επιλογές που έχουμε. Και πρέπει να σας πω ότι καμία επιλογή δεν εξαιρέθηκε. Όμως να πω το εξής. Καταρχήν εμείς θέλουμε να υπάρχει θετική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε ή δυνατόν. Και δεύτερον, έχω καταστήσει σαφές τις συζητήσεις μου με την ε, κυβέρνηση και τον πρόεδρο ότι ανησυχούμε πάρα πολύ και ότι εξετάζουμε όλες μας τις εναλλακτικές λύσεις. Και νομίζω ότι το μήνυμά μου έγινε κατανοητό. Για την κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία ε, θα πρέπει σύντομα να φτάσει τόπου η αποστολή μας και το θέμα δεν είναι να φτάσει η αποστολή βεβαίως μετά τη γενοκτονία. Η εφαρμογή, η πλήρης ανάπτυξη μιας αποστολής από το δικό μας το πρίσμα δεν είναι κάτι το απλό, σαν να έχει δηλαδή κανείς ε, στρατιωτικές δυνάμεις στη διάθεσή του περνώντας τα χρόνια και νομίζω όλοι το έχουμε κατανοήσει καλύτερα το πώς μπορούμε να λειτουργούμε και το τι μπορούμε να κάνουμε. Το να υπάρχει ε, μία ομάδα ταχείας αντίδρασης με σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ίσως να μην φτάσουμε και ποτέ. Πάντως τώρα δεν είμαστε ακόμα εκεί. Γι' αυτό λοιπόν ε, αναζητούμε κράτη-μέλη ε, για να βοηθήσουν όσο καλύτερα μπορούν και να μπορούμε κι εμείς ε, να στηρίζουμε με αποστολές επιτόπου. Αυτό που έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά είναι να κάνουν οι αποστολές αυτές αυτό που τους λέμε να κάνουν και να παραμένουν μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ ακριβώς γιατί παραμένουμε επί τόπου ε, όπου πάμε, ας πούμε στην περίπτωση της πειρατείας, εκεί ε, το 95% της αποστολής εκπληρώθηκε. Η δουλειά που κάνουμε είναι πραγματικά σημαντική. Ε, ο αρμόδιος διοικητής έχει μεταβεί στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία αυτή την εβδομάδα. Θα δω βέβαια τις πληροφορίες. Αυτό που έχει βέβαια μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η αρμόδια επιτροπή ε, θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως. Και σχετικά με την ερώτηση του κ. Ντανζόν, πράγματι αρκετά κρατημέλη έχουν προτείνει να συμμετάσχουν σε αυτή την αποστολή. Τώρα, για τη Λιβύη, ε, πολλά κρατημέλη δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν Τώρα λοιπόν προσπαθούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τους συνεργάτες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να προχωρήσουμε όχι μόνο στο θέμα της ασφάλειας αλλά και των θεσμών. Γιατί πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Λιβύη οφείλονται στο ότι δεν υπάρχουν οι θεσμοί όσον αφορά την ασφάλεια, βεβαίως η κατάσταση επιδεινώνεται. Και όταν ο Πρωθυπουργό δεν μπορεί να προσγειωθεί στην πατρίδα του, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Κατά την άποψή μου, ο συντονισμό είναι πάντα απαραίτητο και χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό. Όσον αφορά τη Συρία, ξέρετε, δεν υπήρξαν ακόμα συμπεράσματα γιατί ε, δεν έχει υπάρξει πρόοδος, έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ανταυτού να έχουμε συζήτηση. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και μια σωστή επιλογή. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Απλά υπάρχει το αίσθημα ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να προχωρήσουμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένοι και μου, συναντηθήκαμε με στελέχη της αντιπολίτευσης ε, στη Συρία, ε, και στον κόλπο που πήγα πρόσφατα και προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση. Στη Γενέβη 2 ε, καθόμουνα δίπλα σε έναν κύριο από ένα καθεστώς ε, εκεί της περιοχής και είχαμε μία μακροσκελέστατη συζήτηση. Πάντως πρέπει να προχωρήσει πράγματι η ε, συζήτηση και να υπάρξει και σχετική συμφωνία. Κύριε Σουβελόφ, ο κύριος Σουβελόφ, ο αναπληρωτής Όσο μιλάει για την Τελωνιακή Ένωση, υποτίθεται ότι θα ε, ξεκινήσει το Μάιο ε, και αυτό έχει ως στόχο να επιτευχθεί η Τελωνιακή Ένωση στην οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένο ο κύριος Πούτιν και θα δούμε πώς προχωράει. Βεβαίως ε, θα παρακολουθούμε την κατάσταση και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με τη Ρωσία για το θέμα αυτό. Για την Ουκρανία νομίζω ήδη απάντησα για το θέμα των κυρώσεων και για το τι είπε η Βικτόρια. Μια άλλη ερώτηση κατά πόσον και οι δύο πλευρές μας αντιμετωπίζουν ως διαμεσολαβητή στην Ουκρανία. Ξαρτάται πώς ορίζεται το διαμεσολαβητή. Αυτό που ισχύει είναι ότι έχουμε πρόσβαση και στις δύο πλευρές. Εγώ συναντήθηκα με τον πρόεδρο και στις δύο φορές που πήγα. Είχε τη διάθεση να συναντηθεί μαζί μου και συναντήθηκα και με όλα τα στελέχη της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία. Και πρόσφατα συναντήθηκα μαζί τους και στο Μόναχο. Τους προσφέραμε λοιπόν ε, την υποστήριξη που κρίνουν εκείνοι ότι θα τους βοηθήσουν βοηθήσει καλύτερα. Και θέλω να σας πω ότι δεν έχει νόημα να πάρουμε έναν ειδικό εμπειρογνώμονα για τα συνταγματικά οτιδήποτε άλλο. Ε, ό,τι θέλουν μπορούμε να τους προσφέρουμε, αλλά εκείνοι πρέπει να το ορίσουν και εμείς έχουμε ήδη προτείνει, θα δούμε κατά πόσον θα δεχτούν την προσφορά μας ή όχι. Κατά πόσον στη συνεργασία με την Ουκρανία έχουμε πει την τελευταία μας λέξη, κοιτάξτε, ο στόχος δεν είναι η συμφωνία γιατί μπορούν ε, να υπάρξουν πολλές ερμηνείες για το πού θα προχωρήσει το μέλλον η συνεργασία με την Ουκρανία. Και βεβαίως και τα κράτη-μέλη μπορεί να έχει το καθένα τη δική του ερμηνεία. Όμως αυτό που ε, συμφωνούν όλοι είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί και να εμβαθυνθεί η σχέση και πέρα από τη συμφωνία. Τώρα για την Βοσνία, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλο αυτό δεν θα εξελιχθεί σε σύγκρουση και ε, σίγουρα όχι για εθνοτικούς λόγους. Νομίζω τώρα πρέπει να παρέμβουμε, γιατί ακόμα και στις συγκρούσεις που είδαμε πρόσφατα βλέπουμε να υπάρχουν κάποια στοιχεία που ε, θα ήθελαν να μετατοπίσουν τη σύγκρουση αντί να είναι για οικονομικά θέματα να είναι για άλλα θέματα. Σε Ρόμπερτ σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ για τα σχόλιά σας ε, σας ευχαριστώ, το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό που είπατε για μένα. Τώρα, για την Μέση Ανατολή. Νομίζω ο κύριος Κέρι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έδειξε ιδιαίτερη στράτευση για αυτό το θέμα, είναι απόλυτα αποφασισμένος, μιλάω πολύ συχνά μαζί του για όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει και θα συνεχίσει να εργάζεται επί του θέματος αυτού, γιατί είναι μία από τις πρώτες του προτεραιότητες. Υπάρχει μεγάλη ε, στράτευση ε, και επαφές με το Ισραήλ, ένα πλαίσιο θέλει να καθορίσει ο Σύπνε Λίβνη είναι ο ε, επικεφαλής των, ή επικεφαλής των ε, διαμεσολαβητών από πλευράς του Ισραήλ. Γνωρίζω και αυτή την πλευρά και των Παλαιστινίων. Ξέρω ότι ε, προχωράνε καλά. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Νομίζω λοιπόν υπάρχουν κάποια ε, στοιχεία πρόοδου. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση συνασπισμού υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Αυτό που είναι ε, σαφές είναι ότι στο Ισραήλ πολλοί πιστεύουν ότι αν υπάρχουν τα σωστά εχέγγυα για την ασφάλεια και ουσιαστική κατανόηση του μέλλοντος του Ισραήλ τότε καλύτερα να υπάρξει συμφωνία από το να μην υπάρχει καθόλου. Και νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη του Πρωθυπουργού. Εμείς έχουμε πει ότι θα δώσουμε πρωτόγνωρη βοήθεια και προς τις δύο πλευρές εφόσον καταλήξουμε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Κύριε Μάγερ, εσείς ε, μιλήσατε για παρεμβάσεις. Εμείς ε, δεν παρεμβαίνουμε. Ε, πριν δέκα μέρες, πριν από τη συνάντηση κορυφής, πρόκειτο το, τη μονογραφημένη συμφωνία να την υπογράψουν ομόφωνα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρόβλημα. Μας είπαν ότι το πρόβλημα ήταν οικονομικής φύσεως για βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Πήγα λοιπόν επιτόπου για να μιλήσω για αυτές τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και στις επισκέψεις που έκανα ε, μίλησα με όλους και καταστήσαμε σαφές ότι εμείς δεν είμαστε για να παρεμβαίνουμε αδικαιολόγητα, οποτεδήποτε όμως προκύπτει ε, βία, εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε στο να εξευρεθεί συμφωνία. Εκεί φέρουμε κάποια ευθύνη. Δεν είναι ότι ε, μπερδευόμαστε χωρίς να μας θέλουν, θέλουμε να βοηθήσουμε. Το είπα όμως αυτό και στην Ουκρανία. Η λύση ήταν της Ουκρανίας, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνοι πρέπει να αποφασίσουν. Ε, και τους είπα μάλιστα, μην σκέφτεστε σχέδια διαφορετικά κατόπιν τούτου τους καλούμε να προχωρήσουν το διάλογο γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Όμως να είναι ουκρανικό το σχέδιο. Κύριε Ντανζόν, όπως σας είπα... Η δύναμη επιχειρήσεων στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι έτοιμη. Η Εστονία έχει ε, εγγύηθει για την υποστήριξή σας. Είναι 7 κράτη τα οποία έχουν παρουσιάσει επίσης υποσχέσεις για βοήθεια για την ε, δύναμη που θα πάει στην Αφρικανική Επιτροπή. Θα ακολουθήσει μια παρουσίαση στη Στρατιωτική Επιτροπή και στην Πολιτικό Στρατιωτική Επιτροπή για το πώς θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η συνεργασία των ταχυδρομητών. Ελπίζω ότι αυτό θα στεφτεί υπό επιτυχίας. Αναφέρθηκα ήδη στη Λιβύη και αναφέρθηκα και στη Βοσνία. Τώρα θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο, όπως έχουμε σκεφτεί εδώ και πολύ καιρό, για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τη Βοσνία. Προχωρούν όλε οι χώρε της περιοχή, αλλά η Βοσνία υπολείπεται. Όταν μιλάει κανεί με του ηγέτε στη Βοσνία, δεν βλέπει κανείς να υπάρχει μια διάθεση να προχωρήσουν. Πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να του υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος. Συνεχίζουμε με τον επόμενο γύρο. Ένα λεπτό για τους υπόλοιπους. Κυρία Ιμπριζάγκητς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, θα ήθελα να επανέλθω στην ε, ε, Βοσνία, γιατί δεν κατάλαβα πολύ καλά την, ε, την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, δηλαδή πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η αναταραχή που έχει ξεκινήσει δεν θα αποκτήσει εθνοτική χρειά. Ξέρετε ότι στα μέσα ενημέρωσης ε, γράφεται σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις διαμαρτυρίες και ε, προσπαθεί να δώσει εθνοτικό χαρακτήρα και ε, στις, στις καταστάσεις αυτές. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρόκειται για πολύ κεντρικό σημείο και θα ήθελα να καταλάβω καλά την άποψή σας από αυτού. Και ρωτώ λοιπόν πώς προτίθεστε να λύσετε το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω μια ερώτηση που αφορά τη δικιά μου χώρα. Ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας σχετικά με την κατάσταση που σχετίζεται με τους δύο Ιταλούς πεζοναύτες. Είναι παράδοξη η κατάσταση. Ξέρετε ε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, μια ε, διαρκής, ένα κυνηγητό κατά αυτών των ανθρώπων που βεβαίως αποτελεί χαστούκι στην, Ευρώπη, στην Ιταλία και αν μου επιτρέπετε κατ' επέκταση και στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι δεν γνωρίζει μια μεγάλη χώρα ποιες είναι οι αρχές της ειρηνικής αστικής συμβίωσης. Είναι σαφές ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι ε, και επομένως ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει κάποια προσπάθεια έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας κυρία Άστον. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για την Βοσνία. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες διαδηλώσεις γίνονται στην Βοσνιο Κροατική ε, Ομοσπονδία και είναι τα πράγματα ακόμα ήρεμα στη Ρεπουμπλικά Σεύσκα. Και τώρα ο υπουργό της Κροατίας πηγαίνει στο Μόσταρ και ο υπουργό της ε, Ρεπούμπλικα Σέρπκα πηγαίνει στο Βελιδά. Το πρόβλημα βρίσκεται στη συμφωνία του Ντέιτον και έτσι πρέπει να αλωθεί. Εγώ χαίρομαι για την υπομονή του κυρίου Φίλε που λέει ότι θα λυθεί από μόνο το πρόβλημα. 15 χρόνια έχουν περάσει και παραπάνω. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λοιπόν να περιμένουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξέγεση κατά των ε, διοικούντων στη Βοσνία Ζεγοβίνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα. Λέτε ότι χρειάζεται ηγέτε στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Εγώ δεν βλέπω αυτοί οι οποίοι είναι τώρα ηγέτε να παίξουν ηγετικό ρόλο. Θα ήθελα να ξέρω αν πιστεύετε ότι πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε τη συνδίκη της Dayton και να την αλλάξουμε όλοι από κοινού. Κυρία Άστον, ε, φαίνεται ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, βρίσκεται σε ένα σημείο χαμένο ε, στη σφαίρα των, της έλλειψης ενδιαφέροντος και των τοπικών αρχόντων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ανάμεσα στις Βρυξέλλες, την ε, Πρίστινα και την ε, Σερβία γίνονται συζητήσεις, καταφέρνουμε να βρούμε συνολικές λύσεις, αλλά όταν μιλάμε για συμφωνία ανάμεσα στο Σαράβιο και στην Πάνια Λούκα, τελικά δεν καταφέρνουμε να βρούμε συμφωνίες τήρηση των συμφωνιών του Ντέιτον είναι πάρα πολύ σημαντική για την Βοσνία Ζεγοβίνη. Όχι μονάχα για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, αλλά και ώστε η χώρα αυτή η οποία έχει περάσει μέσα από τόσες ταλαιπωρίες να μπορέσει να ζήσει φυσιολογικά. Ε, θα έπρεπε λοιπόν για τη χώρα αυτή να έχουμε ένα γρήγορο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα fast track, έτσι ώστε να εξηγιανθεί αμέσως η κατάσταση στη χώρα αυτή που ταλανίζεται. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θέσω και πάλι το ερώτημα για την περίπτωση Μαγνίσκη στην ε, Ρωσία. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή μας συζήτησε τη νέα αυτή σύσταση προς το Συμβούλιο όπου αναφέρονται και 32 ονόματα για τα οποία θέλουμε να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον τους από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορισμοί για τις ε, βίζες. Θα ήθελα να ρωτήσω τι έγινε με την προηγούμενη σύστασή μας του 2012 που ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν δόθηκε συνέχεια μέχρι τη στιγμή και δεν πήγε στην μέση διαταξή του Συμβουλίου αυτή η σύσταση. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να εγκρίνει μια νέα σύσταση. Πότε περιμένετε ότι το θέμα αυτό θα μπει στην μέση διαταξή του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Κυρία Αστόν, το 2008 είδαμε στη σκιά των Ολυμπιακών Αγώνων να υπάρξει μια επέμβαση των ρωσικών δυνάμεων στην Νότια Οσετία μέχρι και τη Γεωργία. Πολλοί φοβούνται ότι η Ολυμπιακή ειρήνη του Σότσι είναι απατηλή αυτή τη στιγμή. Εδώ και εβδομάδες ακούμε από τον κύριο Μπόγκος και από τον κύριο Γκλάζεφ ότι θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία στην πλατεία Μαϊντάν. Εγώ έχω ακούσει πολύ ανησυχητικά νέα από την αντιπολίτευση της Ουκρανίας που λένε όλο και περισσότερο εμφανίζονται ε, στρατιωτικοί Ρώσοι με στολές ε, ουκρανικές και είναι ένα είδος υφέρπουσας εισβολή στην ε, Ουκρανία. Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το επιβεβαιώσετε μπορούμε να ξέρουμε αν όταν πηγαίνουμε εκεί πέρα παρακολουθούμαστε και εμείς και τα τηλέφωνά μας ή όχι. Φανόρντεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Κύριε Άστον, πιστεύω ότι έχουμε μάθει το δίδαγμα από την τελευταία μας παρόμοια παρέμβαση στην Τσάντ το 2009. Θυμάστε ότι αυτή η αποστολή λειτουργήσε με πολλές δυσκολίες επιμελητίας και άλλες από την αρχή. Αναρωτιέμαι αν πιστεύετε ότι η Αφρικανική Ένωση θα είναι έτοιμη να αναλάβει σκητάλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έξι μήνες. Δεύτερον, βλέπω ότι αναφερθήκατε στα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης του, της τρομοκρατίας. Χαίρομαι για αυτά τα στενάρα μέτρα, αλλά έχετε κάνει κάποια ε, προσπάθεια να καταγράψετε ομάδες που συνδέονται με την Αλκάιντα στην Συρία που στραστηριοποιούνται εκεί και ένα ακόμα σημείο που είναι στην μέση διαταξή σας και το οποίο όμως θα μπορούσε να είναι το θέμα της Ζιμπάμπουε. 20 Φεβρουαρίου ελπίζουμε ότι θα αρθούν τα τελευταία περιοριστικά μέτρα εκεί πέραν αυτών που αφορούν τον Μουγκάμπε. Πιστεύετε ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε να μπορέσετε να άρετε όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα που όπως έχετε ανακοινώσει. Thank you, Mr. Chairman. Last... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα στην, Ομόλια, στην Ολομέλεια ε, ψηφίσαμε έξι ψηφίσματα ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια και την ενταξιακή τους πορεία. Δύο θέματα η συμφωνία με το Κωσυφοπαίδιο και τη Σερβία. Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δείξατε ότι η, διπλωματία είναι η τέχνη του ανέφικτου. Ε, μάλλον της επίτευξης αυτών που αρχικά φαίνονται ανέφικτα. Ε, πιστεύουμε ότι τέτοιες συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν τη σταθερότητα ε, στην περιοχή. Βοσνία Ρεζεγοβίνη τώρα. Όλοι ε, αναρωτιούνται τι θα γίνει με την κατέσταση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα πολύ αυστηρό ε, πρόγραμμα το οποίο θα συμφωνηθεί από όλες τις χώρες, από κάθε μία από τις χώρες και όχι όποτε θέλει η μία. Λυπούμε, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και οι χώρες να είναι εξαιρετικά πειθαρχημένες. Οπωσδήποτε να ε, γίνει αυτή η συμφωνία. Απάντηση. Κυρία Μπριτσικτσικ. Δεν το πρόφερα και πολύ καλά. Ας την πούμε Άννα καλύτερα. Αγαπητή Άννα λοιπόν. Είναι σοκαριστικό να σκέφτεται κανείς, ε, ε, ακόμη και να σκεφτεί κάποιος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πίσω από αυτές τις ε, ταραχές στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Με σοκάρει και μόνο το ενδεχόμενο αυτής της σκέψης. Υπάρχουν δύο-τρία στοιχεία τα οποία πρέπει να γνωρίζει κανείς. Πρώτον, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία ε, στο Σαράγεβο και σε άλλες περιοχές έχουν δώσει δείγματα ε, ιδιαίτερης ε, κατάστασης. Ε, υπάρχουν, υπήρχαν κάποια πρόδρομα σημάδια. Ε, και εμείς ε, βεβαίως ε, από την δικιά μας πλευρά στείλαμε συγκεκριμένα μηνύματα προς όλους τους ηγέτες ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή και να μένετε με σταυρωμένα χέρια, πρέπει να κάνετε κάτι. Κατεβλήθησαν πολλές προσπάθειες και θα θυμάστε ότι λίγο πριν λήξει η θητεία της Χίλερη Κλίντον είχαμε επισκεφτεί την περιοχή. Θυμάμαι ότι αισθανθήκαμε μεγάλη αγωνία προσπαθώντας να στηρίξουμε την Βοσνία Ζεγοβίνη έτσι ώστε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυτή ήταν η δικιά της ε, ε, σκέψη, αλλά και για να συνεχιστεί ο διάλογο. Θέλαμε να του δείξουμε ότι στην ουσία μπορούσαμε να βοηθήσουμε ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και οι Ηνωμένε Πολιτείε, μπορούσαμε να βοηθήσουμε με πολλαπλού τρόπου. Νομίζω ότι τα μηνύματα αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να επαναλάβουμε. Έκτοτε έγιναν πολλά, πολλά πράγματα και οπωσδήποτε ε, και όλη η ομάδα της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης έχει, ε, έχει δουλέψει πάρα πολύ επί τόπου. Είχαμε επανειλημμένες επισκέψεις. Τώρα, πριν τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου ε, είχαμε αναφέρει και το ζήτημα της Βοσνίας Αζεγοβίνης λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια περιφερειακή προσέγγιση. Ε, επιματέω όλα αυτά. Η κατάσταση σήμερα ε, από οικονομικής απόψεως τουλάχιστον ε, ακόμα είναι σε πολύ, ε, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο κόσμος είναι εξαιρετικά αγχωμένος με όλη αυτή την, την κατάσταση και Επομένως ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να μπουν και τα οικονομικά σε μια σειρά και να ακολουθήσουν και τα πολιτικά. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς ε, τέτοιες ε, λύσεις. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συζητούμε μαζί τους έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν ποια είναι η κατάσταση. το πρόβλημα και έχετε δίκιο ότι υπήρχαν κάποια σημάδια όσον αφορά την, ε, την εθνοτική διάσταση και στο Σαράγεβο και το Μόστρα που το παρακολούθησε και από πιο κοντά. Ε, υπήρχαν κάποια πρόδρομα σημάδια αλλά, και νομίζω ότι ε, πρέπει να είμαστε πιο παρόντες. Η παρουσία μας θα πρέπει για μία ακόμα φορά να είναι πιο έντονη επιτόπου. Ε, μίλησα και με τον Σέρβο και με τον ε, Κροάτι και με τον Τούρκο ε, Πρωθυπουργό ή με Υπουργό Εξωτερικών έτσι ώστε να δούμε κοινό τρόπο δράσης. Όσον αφορά κύριε Παντζέρη αυτό που ρωτήσατε για τους Ιταλούς πεζοναύτες όχι μονάχα μας προβληματίζει ιδιαίτερα, δηλαδή όχι μόνο είναι ε, πολύ κακό για την Ιταλική κυβέρνηση, αλλά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Εάν ε, ληφθεί ε, μια απόφαση και εάν θεωρηθούν ε, ότι ε, η δράση των Ιταλών πεζοναυτών στα πλαίσια μιας αποστολής καταπολέμησης της πειρατείας, εάν θεωρηθούν, λέω, ε, ενταχθούν στον αντιτρομοκρατικό νόμο, τότε οπωσδήποτε θα μας βρουν αντιμέτωπους. Έχουμε ήδη στείλει επανειλημμένα το μήνυμα, έχουμε κάνει διαβήματα και προφορικά και γραπτά, επανειλημμένα έχουμε συζητήσει και με τον ε, σύμβουλο του Εθνικού Συμβουλίου ε, και μάλιστα το συζητήσαμε και προημερών με αυτό. Δεν είναι το ζήτημα αν θα ε, υπάρχει θανατική ποινή, μάλλον δεν θα υπάρξει θανατική ποινή, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο οι δύο πεζοναύτες να δικαστούν με απαγγελία κατηγοριών υπό τον αντιτρομοκρατικό νόμο και βεβαίω θα συνεχίσουμε ε, να, σε συνεργασία και με τους ε, Ιταλούς συναδέλφους ε, να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Κυρία Πακ. Αναφερθήκατε ε, στο ε, ζήτημα ε, του ότι πρέπει να κινηθούμε προς κάθε κατεύθυνση. Σας είπα ότι και χθε μίλησα με τον, Ιταλό, συγγνώμη, με τον Τούρκο, με τον Κροάτη, αρμόδιο υπουργό. Βεβαίως είναι πολλές οι χώρες οι οποίες στηρίζουν την Βοσνία Ζεγοβίνη ο Πρωθυπουργό και ο αναπληρωτής Πρωθυπουργό και της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου ε, θα ε, είναι παρόντες ε, στην 21η, αν δεν κάνω λάθο συνεδρία του διαλόγου που έχουμε ξεκινήσει και βεβαίω το πρώτο σημείο στη μέρη σε διάταξη είναι η Βοσνία Ζεγοβίνη. Είπα ότι πρέπει να υπάρχει περιφερειακή συμφωνία. Ε, βεβαίως ε, το ε, ένα μοντέλο δεν μπορεί να ισχύσει για όλες τις περιοχές. Θα πρέπει με τον πλέον δόκιμο τρόπο να λύνονται τα περιφερειακά προβλήματα. Απλώς είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγκάρσια συνεργασία διακοινοτική, διεθνοτική. Again, I've mentioned Κύριε Πίτσουλα. Ε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και είναι γεγονός όπως πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει το κομμάτι που φαίνεται και υπάρχουν και όλα τα ζητήματα τα οποία ε, αφορούν την πολιτική και οικονομική αποτελμάτωση της χώρας. Ε, βλέπουμε πώς είναι η ζωή, υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν είναι αθρηρή η οικονομία, δεν υπάρχει, υπάρχει μάλλον πρόβλημα ε, πολιτικής ε, ηγεσίας. Υπάρχουν γενικά προβλήματα κινητηρίων δυνάμεων που θα οδηγήσουν τη χώρα προς τα εμπρός. Ε, και επειδή μόνοι τους προφανώς δεν θα μπορέσουν να, βρουν, τη λύση, οπωσδήποτε θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς. Αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Η κυρία Όγιουλαντ με ρώτησε για την υπόθεση Μαγνίτσκι. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πρωτοφανή βήματα. Ε, έχουμε διαβήματα, έχουμε δηλώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου. Αυτή η μεταθάνατον ε, καταδίκη ε, έχει αναφερθεί σε όλες τις διαβουλεύσεις που είχαμε με την Ρωσία και στους, στο διάλογο που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδεχομένως δεν γίνεται αναφορά εξπρέσεις βέρμπης κάθε φορά στο ζήτημα αυτό, αλλά οπωσδήποτε ε, ε, το μήνυμα περνάει και επανειλημμένα έχουμε πει πώς πρέπει ε, να αντιμετωπιστεί το, το ζήτημα. Και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει η ρωσική πλευρά. Σχετικά με τη Γεωργία, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Πάντως, εγώ δεν έχω ακούσει να υπάρχουν τόσοι πολλοί Ρώσοι σύμβουλοι στην Ουκρανία. Εγώ δεν είδα κανέναν. Αλλά εντάξει δεν έπρεπε και απαραίτητα να το ξέρω. Πάντως κάπου έχετε δίκιο. Κυκλοφορεί το ότι οι Ρώσοι προσφέρουν υποστήριξη. Ε, θα ισχυριστούν βέβαια οι ίδιοι ότι κάνουν και αυτοί ακριβώς το ίδιο, προσφέρουν υποστήριξη σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίση. Όσον αφορά τις ε, στολές ε, που φορούν, νομίζω ότι και οι δυο μας γνωρίζουμε την απάντηση επί του θέματος. Κύριε Βανόρντεν, σχετικά με την κεντρική αφρικανική δημοκρατία, νομίζω ότι έχουμε μάθει το μάθημά μας, γιατί σε πάρα πολλά κράτη Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει κανείς ε, κάπως να τα στηρίξει και ένα πράγμα που είναι καλό είναι ότι η στρατιωτική συνεργασία δεν ξέρω αν έχετε πάει στο βαράκι που είναι η αποστολή Αταλάντα ο διοικητής και οι προκάτοχοί του ανέκαθαν έλεγαν ότι ένα πολύ καλό πράγμα στη συνεργασία είναι ότι έχει κανείς πάντα κάτι να μάθει, εμπειρία και γνώσεις και αυτό βοηθάει το να βελτιώνεται σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης και άλλα παρεμφερή. Η Αφρικανική Ένωση έχει ήδη ε, αναλάβει, έχει ήδη στείλει δυνάμεις επιτόπου στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και τώρα το ε, Σεπτέμβρη θα στείλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα Ηνωμένα Έθνη αποστολή. Ξέρουμε ότι υπάρχει σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, όσον αφορά... Ξέρετε πόσο σοβαρά λαμβάνουμε διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται για τη Συμπάμπουε. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με τη διαδικασία. Νομίζω η απάντηση στην ερώτησή είναι ότι πράγματι και εμείς αυτό πιστεύουμε. Δηλαδή, όχι μόνο υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη, το ξέρετε εσείς αυτό καλύτερα, αλλά υπήρξαν επίσης συζητήσεις και με πάρα πολλούς ε, πολιτικούς επιτόπου, τους οποίους εγώ έχω συναντήσει πολλούς εξ αυτών οποτεδήποτε έρχονται στις Βρυξέλλες. Νομίζω λοιπόν ότι σωστά πράττουμε τώρα. Στην περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση θα μπορέσουμε να αποσυρθούμε, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η στιγμή και έχω την αίσθηση ότι στη Ζιμπάμπουε κάπως προχωρούν ε, τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι προχωράει η κατάσταση και πρέπει να την παρακολουθήσουμε εκ του σύνοικης. Ο κύριος Κούκαν σχετικά με τη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο. Κοιτάξτε, με τις συζητήσεις πετύχαμε πολλά. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε και στη Βοσνία, γιατί αυτό είναι αντίφαση. Στη Βοσνία η ηγεσία πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει. Να συνειδητοποιήσουν ότι για να προχωρήσει η χώρα πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Και αυτό είναι καθαρά δική τους απόφαση. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα ένα γύρο τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κύριε Λίζεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μίλησε στα σουηδικά κύριε Μπραζίγκητς, εγώ θα μιλήσω πολωνικά. Ε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της γεωργίας εν συντομία. Γιατί είμαι εισηγητής για το θέμα της γεωργίας. Ο κύριος Σούλτς αναφέρει και στο ζήτημα αυτό. Αλλά πρόκειται για την ε, δημιουργία μιας ζώνης ε, ασφαλείας στην Απχαζία στην περίπτωση των Ολυμπιακών του Σότσι. Στο τελευταίο μας ψήφισμα από το Στρασβούργο το τονίζουμε ότι υπήρξε μια δημιουργία άτυπων συνόρων στην Γεωργία. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες υποδομές στο εσωτερικό της Γεωργίας και έχει συνεχιστεί αυτό το θέμα μέσα στην περιοχή που ελέγχουν τα ρωσικά στρατέματα. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και πώς θα τη σταματήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άστον, ένα βαρονέσα Άστον, ένα ερώτημα για την Συρία. Τα χημικά όπλα υποτίθεται ότι έχουν ε, καταστραφεί, αλλά συνεχίζεται ο πόλεμος. Πεθαίνουν τα παιδιά, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν πια φάρμακα. Πώς προχωράει λοιπόν η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η αθλειότητα και τα βάσανα των ε, προσφύγων. Και ανεξάρτητα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες εξακολουθούν να υπάρχουν επαφές με την ε, Ρωσία ή τα έχουμε θαύσει στο, στο Ολυμπιακό χιόνι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε λοιπόν την κατάσταση των ε, προσφύγων, ακόμα και, με τα, και χωρίς χημικά όπλα μπορούν να πεθάνουν οι άνθρωποι με φρικτό τρόπο και η τύχη των παιδιών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Ευχαριστώ. Από τους Βρετανούς συντηρητικούς δεν θα σας ρωτήσω πού ακριβώς θα πατήσει κανείς όταν πατάει σε ευαίσθητα σημεία της ε, Συρίας. Εγώ άκουσα για... την Ουκρανία, τη θέση του... της Ουκρανίας δεν βλέπω το Συμβούλιο να έχει πει κάτι και προφανώς η ρωσική ε, συμμετοχή είναι πάρα πολύ κέρια για την επιτυχία της συνδιάσκεψης Γενέβη 2. Μπορείτε να μας πείτε κάτι σε σχέση με τις δυνατότητε η Ρωσία να αναλάβει ένα πιο επικοδομητικό ρόλο για την επίλυση της κρίσεως της Συρίας. Ο κύριος Ποπόσκι από την ε, Πουδογομού ήταν ε, παρόν σε ένα δείπνο εδώ χθες. Εγώ προσπαθώ να αναχαιτήσω τις αντιπαραθέσεις που γίνονται εκεί. Είχα συζητήσει με τους Έλληνες για το τι μπορούν να πετύχουν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια για το πώς έχει προχωρήσει το Συμβούλιο με αυτή την υποψήφια χώρα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Άστον, ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι εσείς παίξετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη σχέση μας με την Ελβετία και την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων μετά το δημοψήφισμα. Το ερώτημά μου είναι θα πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλήσατε χθε με τους συναδέλφους σας για το ταξίδι αυτό. Τι περιμένετε από τη διασκέψη κορυφής που θα γίνει την, τον επόμενο μήνα με τον πρόεδρο Ομπάμα στις Βρυξέλλες το Μάρτιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ο κύριος Ιζετμπέργκοβιτς από την κυβέρνηση της Βοσνίας Εζεγοβίνης λέει ότι όλη αυτή την κρίση θα την αντιμετωπίσει σε σταθερή επαφή με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Αν η Τουρκία θέλει να δώσει βοήθεια για τα θέματα αυτά, πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί με αυτά που είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρατήσει ένα ηγετικό ρόλο. Ο κύριος Ιζετμπέκοβιτς ήταν μαζί σας σε επαφή με κάποιους άλλους ηγέτες της ε, Βοσνίας και ποια συγκεκριμένα διπλωματικά βήματα θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Σας. Ευχαριστώ κυρία Άστον. Ε, συγχαρητήρια και για την ε, υποψηφιότητά σας για βραβείο Νόμπελ. Ε, μαθαίνω με ευχαρίστηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάτε στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι Κούκαν και η Μπρεγιά Γεζεβίτς ε, κάποιες ε, λύσεις από τη στιγμή που ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια τους πολιτικούς και από τη στιγμή που οι χώρες είναι διστακτικές θα πρέπει να επιβληθούν ο κόσμος, ο οποίος έχει βαρεθεί πλέον και δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς, ε, ε, ευελπιστεί, προσδοκά ότι εσείς ε, σαν εκπρόσωπος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρετε κάποια, ένωση, κάποια λύση. Δεν θέλουμε καμία λύση πασαρέλα, δεν θέλουμε καμία λύση η οποία... years. time, meantime, δεν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ε, ε, πρέπει να λειτουργήσει η χώρα κανονικά. Αυτό περιμένουν ε, και οι πολίτες και θα πρέπει οπωσδήποτε να πιέσετε ή να βοηθήσετε τους ντόπιου πολιτικούς έτσι ώστε να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, πώς βλέπετε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, την, ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν από κοινού σχέδια για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ουκρανία. Επίσης θα ήθελα να ξέρω σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα αν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος με την Ουκρανία. Είχαμε ήδη υπογράψει μια συμφωνία, αλλά ε, η Ουκρανία μας έχει απογοητεύσει σε σχέση με τον αγωγό South Stream και δεν θα έχουμε ουσιαστικά συνεργασία για το θέμα αυτό. Ίσως λοιπόν η Ουκρανία θέλει να βγει από την ενεργειακή συνεργασία μαζί μας. Πώς το σχολιάζετε. Δύο σύντομα ερωτήματα κυρία Άστον. Πρώτα απ' όλα πότε περιμένετε από τις διαπραγματεύσεις μας με τις ΗΠΑ και τον Καναδά να υπάρξει μια λύση των προβλημάτων για τις προξενικές θεωρήσεις με ίση μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρετε ότι υπάρχουν πέντε κράτη-μέλη που έχουν ακόμα την υποχρέωση προξενική θεώρηση για να μπουν στι ΗΠΑ, στον Καναδά και σε άλλε χώρε. Ένα δεύτερο ερώτημα πιο οργανωτικού χαρακτήρα μα απασχολεί πάρα πολύ οι, α, οι ε, για την παρουσία διπλωματών από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες που είχαν συνδεθεί με τι μυστικέ υπηρεσίε των χωρών του στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχετε τέτοιους υπαλλήλους ή κάνετε κάποιο έλεγχο σχετικά. Ναι. θέλετε να απαντήσετε, λέει ο πρόεδρος. Κύριος Καζάκ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπατή, εκπρόσωπε, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στο Ιράκ αναφέρατε ότι η βία αυξάνεται στο Ιράκ και πριν από λίγο καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε ένα ψήφισμα σε σχέση με την ολέτρια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μειονότητες, κυρίως η μειονότητα του Τουρκουμενιστάν ε, στο Ιράκ. Βλέπουμε κάθε μέρα να γίνονται επιδρομές, οι άνθρωποι δολοφονούνται απλά επειδή ζουν στο Κερπούκ που είναι μια περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται τόσο οι Κούρδοι όσο και οι Ιρακινοί. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει αρκετά για να προστατεύσει αυτή την μειονότητα. Εσείς τι πιστεύετε μπορεί να γίνει κάτι για να διευκολυνθεί η κατάσταση. Ο κύριος Πλένκοβιτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι ε, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε σχετικά με τη Βοσνία Ερσεγοβίνη και πρέπει όλοι να προσέξουμε ε, να μην ε, βλέπουμε μόνο αυτή την διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, γιατί σε τελική ανάλυση ε, έγινε η διάρρηξη αυτή υπήρξε στο σύνολο της επικράτειας της χώρας. Ο κύριος Σόνεσον, ο κύριος Ιψκο και πάρα πολλοί άλλοι ε, παρακολούθησα τι ακριβώς γίνεται και τη δική σας την επίσκεψη τη Δευτέρα. Πρέπει να ε, δράσουμε ταχύτατα, να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Η Βοσνία Ερσοκοπίνη να παραμείνει κοντά μας, γιατί δεν νομίζω ότι δικαιούμεθα να υποπέσουμε και πάλι σε ένα δεύτερο ιστορικό λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι ε, είπατε ότι αυτές ε, οι, ε, αυτές οι αναταραχές οφείλονται στην οικονομική και κοινωνική δυσπραγία, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να στείλουμε και κάποια μηνύματα. Εμείς, οι Κροάτες, ανησυχούμε ιδιαίτερως για την κατάσταση στην Βοσνία Ριζεγοβίνη και πρέπει να ανησυχεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή η χώρα έχει χίλια χιλιόμετρα εξωτερικών εξωτερικά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει να βρεθεί οποιοδήποτε κάποια λύση. Ερώτηση λοιπόν, με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε στην επίλυση αυτής της κατάστασης και να βελτιώσετε γενικότερα την ε, κατάσταση που ισχύει στη χώρα αυτή. Σας ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Με κάθε σεβασμό προς αυτά που λέχτησαν μέχρι τώρα σε σχέση με τη Βοσνία Ερσεγοβίνη, επιτρέψτε μου και εμένα να πω το εξής. Βεβαίως και σας σέβομαι, όπως και το χρόνο μας και θα είμαι σύντομη. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση και δύο ερωτήσεις. Γνωρίζω πολύ καλά την δύσκολη κοινωνική κατάσταση και την απογοήτευση των ανθρώπων. Πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου ότι η αναταραχές που βιώνουμε αυτή τη στιγμή δεν αφορούν μόνο κοινωνικής φύσεως θέματα και έχω δύο ερωτήσεις να υποβάλω. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων από αυτή τη μορφή βίας και πώς μπορούμε να ε, προστατεύσουμε ε, τους Κροάτες ε, που είναι πολυπληθείς στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Και επίσης γνωρίζουμε ότι ορισμένες διαδικασίες ταχύτατα μπορούν να προκύψουν από την πίσω πόρτα ενώ προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς διαδραματίζεται στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ξεκινάω με την ερώτηση για τη Γεωργία, για το ρόλο της αστυνομίας ε, και για αυτές τις μετακινήσεις ε, σχετικά με τα σύνορα. Κοιτάξτε, και εγώ ανησυχώ ε, τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή σε σχέση με τις αστυνομικές περιπολίες. Και ξέρω, τουλάχιστον για την κυβέρνηση της Γεωργίας, υπάρχουν κάποιες ε, μετακινήσεις, κάποιες κινήσεις που λαμβάνουν χώρα και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε με την ε, αποστολή που ελέγχει τι ακριβώς ε, συμβαίνει, να συνεχίσουμε να μιλάμε σε κάθε μονομένη περίπτωση για την εδαφική ακαιρεότητα της Γεωργίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπογράψαμε συμφωνία με τη Γεωργία και η Γεωργία αισθάνεται ότι όλοι μας θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να πιέζουμε για την θέσπιση του ψηφίσματος που συμφωνήθηκε, που δεν έχει όμως ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ικανοποιητική λύση για την εδαφική ακαιρεότητα της Γεωργίας. Αυτά τα μηνύματα είναι πολύ σημαντικά. Με ρωτήσατε κατόπιν για τη Συρία, για την ανάγκη να ε, προσφέρουμε φέρουμε υποστήριξη κυρίως ε, στους πρόσφυγες. Μιλάμε για 6,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπιστέντες στη Συρία και όπως ξέρετε υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων που υποφέρουν και μέσα και έξω από τη χώρα. Ξακολουθούμε να είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής ε, το Κουβέιτ τον Ιανουάριο συγκαλέσαμε στην διάσκεψη για να συγκεντρωθούν μεγαλύτερα κονδύλια και τα Ενωμένα Έθνη εξέδωσαν και αυτά έκκληση, αλλά δεν αρκούν τα χρήματα. Δεν αρκούν διότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Το ένα πρόβλημα είναι τα φάρμακα και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γοναριστούν όλα αυτά που είναι απαραίτητα, αλλά και πώς θα φτάσουν εκεί. Καθώς οξύνεται όλο και περισσότερο η κατάσταση, επειδή υπάρχουν διάφορες ομάδες ανθρώπων, είναι δύσκολο να ελέγξει κανείς την κατάπαυση πυρός που προβλέπεται στη διαδικασία Γενέβη 2, αλλά πολύ δύσκολο να μεταφέρει κανείς ε, στη χώρα ε, βασικά φάρμακα, όσο και αν έχουμε αναζητήσει εξελιγμένες λύσεις. Ε, με βάση συμφωνία Γενέβη 2 πρέπει να εξευρεθούν περισσότερα πόροι. Αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και ελπίζω ότι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα δώσουν περισσότερα χρήματα. Και κάτι άλλο να σας πω ότι μας απασχολεί και η ανοικοδόμηση Συρίας όταν θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ε, όσον αφορά τις κυρώσεις, του Συμβουλίου ήταν ε, σιωπηρές αν θέλετε, με την εξή έννοια. Ξέρω ότι στο πλωστάσιό μας έχουμε πάρα πολλά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενώ όμω ότι οι άνθρωποι να προστατεύονται όπου και αν βρίσκονται και να είμαστε σίγουροι ότι προσφέρουμε υποστήριξη. Σε αυτό το πλουστάσιο έχουμε και άλλα εργαλεία που θα τα χρησιμοποιήσουμε αν το κρίνουμε απαραίτητο. Αλλά η γενική μας στάση είναι πάντα να προσπαθούμε να ζητούμε τον επιτυχή διάλογο, να προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους πολίτες και με εκείνους που πραγματικά ενδιαφέρονται να προχωρήσουν. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι αυτά που συμβαίνουν τώρα όσον αφορά δηλαδή της ε, τις ανατραχές στην Ουκρανία, οι αυτούργοι θα πρέπει να δικαστούν, και πρέπει να το αισθανθούν αυτό οι πολίτες ότι πράγματι αποδίδεται δικαιοσύνη. Αυτή είναι η προσέγγιση μας για να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτό που κυρίως απασχολεί τους ανθρώπους που είναι η άσκηση βίας. Μετά βεβαίως υπάρχει το θέμα της ε, πολιτικής ε, κατεύθυνσης. Η ε, συνεργασία με τους Ρώσους για τη Συρία, κοιτάξτε, το συζητάμε αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη Ρωσία. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τη Ρωσία για το Ιράν. Ο επόμενος γύρος συζητήσεων για το Ιράν είναι την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι εκεί και οι Ρώσοι. Είναι βασικοί εταίροι, όπως και στη διαδικασία για τη Μέση Ανατολή. Έχουμε πολλά καλά παραδείγματα συνεργασίας με τους Ρώσους. Και για τη Συρία πρόκειται και για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την επιτυχία της ε, Συμφωνίας Γενέβη 2. Είδα χτες ε, τον κύριο Ποπόφσκι. Οι συζητήσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κάπως ε, συνεχίζονται με την έννοια ότι υπάρχουν κάποια δείγματα ενδεχόμενης πρόοδου. Δεν θέλω να πω όμως πάρα πολλά, γιατί είναι ένα θέμα όπου όλοι γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητο μπορεί να είναι. Το μόνο που μπορώ να επαναλάβω είναι δέστε λιγάκι το τι θα μπορούσε να συμβεί αν επελύονται τα προβλήματα για τη χώρα αυτή. Και αυτό είναι το μήνυμα που πέρασα και χθε. Ε, κατόπιν, όπως σας είπα θα πάω αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι σε τακτική επαφή μαζί τους και ε, για την συνάντηση κορυφή τώρα συντάσσεται η σε διάταξη. Την Τετάρτη, μάλλον μισχύονται την Πέμπτη, θα επισκεφτώ το Λευκό Οίκο και ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε θα είναι το θεματολόγιο της ε, συνάντησης κορυφή. Σίγουρα τα οικονομικά η εμπορική συμφωνία και κατόπιν συζητήσεις για την εξωτερική πολιτική. Ο συνάδελφος Κέρι και εγώ θα συμμετέχουμε στη συνάντηση κορυφής. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία που έχουμε είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για πάρα πολλά θέματα. Και ελπίζω αυτό να φανεί στη συνάντηση κορυφής. Κύριε Στία, με ρωτήσατε σχετικά με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. η απάντηση είναι δεν ξέρω. Εχθές είδα τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών το πρωί και φάγαμε και μαζί το βράδυ. Το βασικό που συζητήσαμε ήταν η συνεργασία. Ε, μιλάμε συνέχεια με την Τουρκία για τη Βοσνία Ερσεγοβίνη και για τις ε, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να στηρίξουμε τη χώρα. Ε, προφανώς όλες αυτές οι συζητήσεις περικλείουν και την Τουρκία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. σχετικά με την ειρήνη που επιβλήθηκε η ειρήνη, κατά πόσο μερικές φορές πρέπει να επιβάλλουμε την ειρήνη. Κοιτάξτε, ε, έχοντας βιώσει κανείς αυτό τον ε, ολέτριο πόλεμο στα Βαλκάνια, η επιβολή λύσης ήταν καθοριστική γιατί τουλάχιστον θα σταματούσε ο πόλεμος. Όμως δεν είμαι σίγουρη σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει τίποτα για να συγκρίνουμε, δεν ξέρω κατά πόσον πολιτικά οι αιρετοί εκπρόσωποι θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν. Είναι διαφορετική η κατάσταση. Ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας, όπως σας είπα, είναι τέτοιος έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται και να μην τίθεται καν επιτάπητο στο θέμα της ε, βίας. Όποιος ε, έχει επισκεφτεί ε, την περιοχή, θα έχετε δει τα τεράστια, τα ε, μεγάλα αυτά νεκροταφεία με τους τάφους ε, και δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε να επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να τους βοηθήσουμε να επιβάλλουν στον εαυτό τους την ειρήνη. Κατά την άποψή μου αυτό πρέπει να γίνει. Κύριε Κόβατσεφ, με ρωτήσατε σχετικά με το αποτέλεσμα των συζητήσεων, ε, σχετικά με τα κράτη-μέλη ε, για τη σχέση με το Καναδά και τις ΗΠΑ. Συνεχίζεται, δεν έχει τίποτα άλλο ε, να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω και αυτά που λένε οι διπλωμάτες και ξέρω ότι δεν το περιμένετε και εσείς να σας το πω. σχετικά με την, ε, τους Τουρκμένους, τη μειονότητα αυτή στο Ιράκ. Νομίζω έχουμε καταστήσει απόλυτα σαφές ε, στη συνεργασία μας με το Ιράκ, με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Πρωθυπουργό, ότι η προστασία όλων των πολιτών στο Ιράκ είναι καθοριστική σημασίας για τη σχέση που θα έχουμε μαζί τους και για τη συμφωνία σύνδεσης. Είναι ένα πολιτικό στοιχείο αυτή της συμφωνίας. Έτσι λοιπόν αυτά όλα εντάσσονται στο διάλογό μας και οτιδήποτε δείχνει ότι οι μειονότητες δεν τυχάνουν σωστή σωστής μεταχείρισης είναι κάτι που τους το λέμε και ε, περιμένουν και τους λέμε πώς να προστατεύσουν τις μειονότητες. Τώρα, δεν έχω εγώ κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά αν έχετε εσείς κάτι που θέλετε να μου επισημάνετε, παρακαλώ. Ο κύριος Πίνκοβιτς, σχετικά με τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Πράγματι, επί τόπου υπάρχουν πάρα πολλοί που συνεργάζονται μαζί μας. Πρέπει λοιπόν να τους στηρίξουμε. Κατόπιν ετέθησαν δύο ερωτήσεις σχετικά με τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Συμφωνώ μαζί σας ότι ένα πρόβλημα είναι που δεν αντιδρούμε είναι η δυνατότητα επενδύσεων. Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια ιστορία στη Βοσνία Σεγοβίνη για την απογοήτευση που νιώθουν οι θεσμοί και οι άνθρωποι. Συμφωνώ λοιπόν επ' αυτού. Και αυτός είναι ένας από τους τομείς που πρέπει να το ξανασυζητήσουμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε ορισμένα προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ε, πράγματι αυτό μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλουμε να προχωρήσει η διαδικασία για να στηρίξουμε του Φίντσι, να λύσουμε οικονομικά προβλήματα για να ε, υπάρξει κάποια ηγεσία στη χώρα, κάτι που σας ομολογώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο. 10 minutes <laughs> Χαίρομαι που μείνατε 10 λεπτά παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και είναι αναπόφευκτο το ότι πήδηξαμε το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις και γίνεται όλο και πιο δύσκολη κατάσταση λόγω των πολλών θεμάτων που έχουμε στην ε, ημερησία. σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο περαιτέρω σας. Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 5 ξεκινάμε στο 4Q1 τη συνεδρίαση μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης και θα μιλήσουμε με τον Τάμπο Μπέκη, τον πρώην πρόεδρο τη ε, Νότιας Αφρικής για παράνομες χρηματικές ροές από την Αφρική. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να έρθει. Ευχαριστώ.